Ah, okay, good. Ε, good afternoon to all. Καλησπέρα σας. Κυρίως το, την άρξη συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι παρόντες εγκαίρως, όλοι σημαντικοί. Καλώς ήρθατε. Κάποιε ανακοινώσει καταρχά. Αύριο έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τέσσερι υπουργού των οικονομικών της Γερμανίας, Ιρλανδία, της Ιταλίας και των κατοχωρών. Ο Γάλλος υπουργό εχθές μας ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσε να έρθει γιατί εν ώψη της Εθνικής εορτή τη Γαλλίας είχε να επιλύσει κάποια ζητήματα σε συνεργασία με τον Γάλλο Πρόεδρο. Έτσι μας το έγραψε. Θέλει δηλαδή να ξεκινήσει αμέσω μετά τι εργασίε τη κοινοβουλευτική τη Εθνοσυνέλευση ο πρόεδρο. Έχουμε λοιπόν τον Γερμανό Υπουργό, τον νέο Ιρλανδό Υπουργό των Οικονομικών, τον Ιταλό, τον Ολλανδό, εκ των οποίων οι τρει έχουν μακρά εμπειρία. Ο Ιρλανδό είναι καινούριο στη θέση αυτή. Πιστεύω ότι είχαμε όλοι τέτοιε επαφές μαζί τους και στο παρελθόν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την υλοποίηση των προϋποθέσεων και των νέων διατάξεων των διεθνών συμφωνιών, ενώ βεβαίως και της εθνικής της ε, συνυπευθυνότητας των κρατών. Βεβαίως, ερώτα θα έχουμε αύριο. Ο καθένας μας από πέντε λεπτά μπορεί να έχει την ευκαιρία να κάνει τοποθέτηση. Ο καθένας από αυτούς μάλλον θα κάνει μια τοποθέτηση πεντάλεπτη αρχικά και θα ακολουθήσει η ε, η φάση των ερωταποκρίσεων. Σύντομες βέβαια και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε αλλάξει κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα με την ε, ακρόαση της Επιτρόπου Γιώργοβα. Η Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει. Εγώ είχα κάποιες αλλαγές στο προσωπικό μου πρόγραμμα που με ανάγκασαν να μεταβώ στη Γερμανία. Μετά έχουμε το, την επίσκεψη στην Πορτογαλία και στην Κύπρο το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Τα πρακτικά είναι υπό προετοιμασία, θα τα δείτε σύντομα. Με διαφορετικές εμπειρίες πρέπει να πω, γιατί εγώ βλέπω ότι από την Πορτογαλία είχαμε πολύ πιο εκρεμή ζητήματα από διάφορες ε, πολιτικές ε, γραμμές και θέσεις διατυπώθηκαν διαφορετικά ερωτήματα. Στην ε, Κύπρο ήταν περισσότερο εστιασμένα στα θέματα της, ε, των τραπεζών, του τραπεζικού τομέα. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης είχαμε την παράταση της εντολής μας έως το Δεκέμβριο, τελευταία παράταση. Συνολικά δηλαδή θα έχουμε 1,5 χρόνο εργασίας. Το αργότερο το Νοέμβριο ή στο ε, το Δεκέμβριο θα πρέπει να κρίνει η Ολομέλεια στις συνόδους της αντίστοιχα τα ε, πορίσματα των εργασιών μας. Αυτά είχα ως ανακοινώσεις. Σήμερα θα δούμε τις προτάσεις των εκθέσεων και των συστάσεων. Θα τις συζητήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ξεκινώντας τη γραμματεία αλλά και τους δύο εισηγητές, Κόφοκ και Ιέτσεκ. Έχουμε και τις μεταφράσεις σε μεγάλο βαθμό έτοιμες, άρα μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα ο καθένας στη γλώσσα του μεταξύ. Και χωρίς να σας ε, καθυστερήσω άλλο, θα επισημάνω ότι έχουμε αρκετή δουλειά. Κάνει. Ασφαλώς οι ομάδες θα έχουν και συμπληρωματικές προτάσεις. Πολύ σημαντικό για μένα είναι να γίνει αξιολόγηση των εγγράφων, να αξιοποιηθούν τα έγγραφα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και τις ε, ε, αποστολές της fact-finding missions. Και επίσης θεωρώ ότι παρότι έχουμε περιορισμένες εξουσίες ως Επιτροπή Διερεύνησης του Σκανδάλου των Αγραφών ε, του Παναμά, ε, καλό θα είναι να κοιτάξουμε και να αξιολογήσουμε και θέματα αντιμετώπισης, διαθεσιμότητας, άρνησης, προσέλευσης των προσκεκλημένων. Κάποιες άλλες σύντομες παρατηρήσεις, πολύ γρήγορα. Ε, μάλλον χωρίς άλλες παρατηρήσεις, μάλλον θα δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές. Ο κύριος Κόφολτ ξεκινάει, Δέκα λεπτά έκαστος παρακαλώ και μετά η Σκιώδης. Γέπε, έχεις το λόγο παρακαλώ για να κάνεις την πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστούμε γιατί για τα όσα είπατε και συμφωνούμε μαζί σας. Έχουμε το πλαίσιο της δουλειάς της Επιτροπής επίσης τις προϋποθέσεις πρόβασης στα έγγραφα, τα έχουμε συζητήσει. Ευχαριστώ και όλους όσους ήρθαν και θα ήθελα αρχίζοντας να ευχαριστήσω και τη γραμματεία μας που επέδειξαν ε, επαγγελματισμό, βοήθησαν πάρα πολύ στην ε, δουλειά και των ε, δύο εισηγητών. Επίσης ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες για τόσα εγγράφους μας στείλανε κατά τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα όσον αφορά το, σχήμα και τη, τη σύνθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, ε, με μεγάλο ενδιαφέρον προσεγγίζεται η δουλειά μεγάλη συμμετοχή αλλά και επαγγελματικό πνεύμα. Πριν μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες του σχεδίου του κειμένου της εκθεσής μας, για να δούμε σε τι πλαίσιο δουλεύουν. Πρόκειται για Εξεταστική Ερευνητική Επιτροπή. Και κλείθημε να διατυπώσουμε κάποια πραγματικά περιστατικά, κάποια στοιχεία, ε, κάποια συμπεράσματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της ε, Επιτροπής, αυτά τα οποία μας βρουν όλους σύμφωνους και είπαμε ότι έτσι θα συνταχθούν τα κείμενά μας και για να σας πω τώρα επίσης για τη διαδικασία. Όπως ξέρετε, αυτό το οποίο θέλουμε να υπάρχει μια έκθεση ε, σύντομη σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα έχει το συμπέρασμα της Επιτροπής όπως αναφέρθηκε. Στο δεύτερο τμήμα θα έχουμε τις ε, συστάσει μας και στο τρίτο τμήμα θα έχουμε σε παράρτημα την περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων, της δουλειά, των ακροάσεων, των αποστολών, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, στοιχείο και για την τεκμήρωσή μας. Και έχουμε μια διαδικασία επίσης για τροπολογίες, ε, όπως ξέρετε πιεζόμαστε από το χρονικό πλαίσιο και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για αναβολές. Με αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δουλεύουμε οπότε. Σας παρακαλώ να επιδείξετε ευελιξία, να έχετε συμβαστικό πνεύμα όσο γίνεται και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων και δύο συνεισηγητές, θα δουλέψουμε μέσα και μετά την ε, ε, προθεσμία για τροπολογίες και βασικές τροπολογίες. Όλοι έχουμε υπόψη ότι όσο πιο ευρεία είναι η συνέντευξη για τα συμπράσματα τόσο πιο ισχυρό θα είναι το μήνυμα προς τα θεσμικά όργανα, προς τα κράτη-μέλη, και για να δούμε τώρα λίγο το θέμα ουσίας. Έχουμε τα εξή θέματα. Πρώτα-πρώτα φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή, τις ε, εξωχώριες ε, ε, δομές, τους φορολογικούς πάντες που δεν συνεργάζονται και καταλήξαμε στο ότι αυτού του είδους οι εξωχώριες δομές, οντότητες, φυσικά νομικά πρόσωπα μάλλον, είναι πολύ σημαντικά για την διάπραξη των ε, εγκλημάτων, αδικημάτων και επίσης έχουμε την νομοθεσία κατά του ξεπλήματος χρήματος και όλα αυτά ε, εν ώψη κάποιων χωρών υψηλού κινδύνου. Οπότε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συντονισμό στη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Το διπλώσαμε αυτό και από τις μελέτες μας και από αποστολές. Και όσον αφορά τις εθνικές διοικητικές αρχές, για αυτά τα αδικήματα, όλα αυτά θα θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία των συστάσεων όσον αφορά τους ε, ενδιάμεσους, τους μεσάζοντες, πολύ σημαντικό κομμάτι γι' αυτό, γιατί εκεί απέτυχε παταγωδός να νομοθετήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει ένα νομικό πλαίσιο για τον ρόλο, το, τις των ενδιαμέσων, των ε, δικηγόρων, λογιστών, τραπεζών, ελεγκτών, των καταπιστευματούχων τέλο πάντων και όλα αυτά οδηγούν σε ένα σωρό εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνες και διαπιστώνουμε ποινικέ ευθύνε. Και εκμεταλλεύονται οι τελούντες τα δικήματα, τα παραθυράκια δηλαδή της νομοθεσίας. Οπότε, να δούμε τι γίνεται στις χώρες. και κατηγορηματικά καταλήγουμε ότι αυτές οι αθέμητες και παράνομες πρακτικές επηρεάζουν δυσανάλογα τι αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε και να ενεργήσουμε μαζί τους. τρόσοφρα τους καταγγέλλοντες και το ρόλο τους. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά και πάλι να δεικνύουμε ότι επήγει να αναλυθεί δράση σε σχέση και με τους καταγγέλλοντες επίσης. Θεσμική συνεργασία. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει ισχύσει η αρχή αυτή της συνεργασίας όσον αφορά τουλάχιστον το Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και ο Πρόεδρός μας τώρα σε αυτό. Σημαντικό αυτό το συμπέρασμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των φορολογικού χαρακτήρα αδικημάτων. Επίσης, δεν πιστεύουμε για επισκεπτός κακοδιοίκησης, οπότε αυτά έχουν σχέση με το κοινωτικό δίκαιο. είναι θέματα διοικητικής συνεργασίας, θέματα εφαρμογής της οδηγίας κατά του ξεπλήματος, ελλείψεις σε εθνικές νομοθεσίες κατά του ξεπλήματος και οπότε ακριβώς όπως έλεγα διαπιστώσαμε περιπτώσεις κακοδίκησης. Και έχουμε και ένα κείμενο για τις συστάσεις μας, προτείνουμε λύσεις και εδώ έχουμε καλύψει πάρα πολλά που πρότειναν οι ηγητές κατά τη συνεργασία μας. Οπότε και λέμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωδημήλη θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο να δεσμευθούν, να στρατευτούν, να ξοδίσουν ό,τι πόρους χρειάζονται και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύσει αυτή τη παντού και διεθνώς Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αυτή η Financial Intelligence Unit. Αλλά πάντως η διαφάνεια είναι η βάση της χρηστής διοίκησης. Έχουμε κάποια σταστικά στοιχεία σε σχέση με φορολογικούς παραδείσους και φορολογικά δικήματα. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για το τι θα κάνουμε με τους φορολογικούς παραδείσους. Θέλουμε θα πρέπει να σταματήσει να χορηγείται φορολογική αμνηστία. Και έχουμε και την έκθεση τάξη, το αποτέλεσμα εκείνης της Επιτροπής μας. Και είπαμε ότι θα πρέπει να, να έχει περισσότερες δυνατότητες ε, η διοίκηση και τα θεσμικά όργανα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για όλα τα επαγγέλματα, εποπτεία ενδιαμέσων και τραπεζών, καταπολέμηση διεθνώς αυτού του ξεπλήματος και να γίνει και μια συνάντηση κορυφής, να σταματήσουν όλους να γίνονται εγκριτό και άρα να υπάρξει τελικά για αυτή τη διεθνώς δράση όργανο ευρωπαϊκό. Προστασία επίσης των καταγγελόντων Οπότε, εν κατακλείδη. Θεωρώ ότι αυτό το κείμενο είναι καλό. Επιδέχεται όμως με τις τροπολογίες σας περαιτέρω βελτίωση. Παρακαλώ και πάλι όλοι να βοηθήσετε να έχουμε συνετικές λύσεις και έτσι να έχουν όσο είναι περισσότερο ειδικό βάρος οι προτάσεις μας όταν εγκριθούν και περιμένω να συνεχιστεί η θετική μας συνεργασία και περιμένω και τις συστάσεις σας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Κόφουτ, για την επισκόπηση αυτή και για την ε, σαφή βούληση για συνενετικές λύσεις. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσουμε να πιέσουμε κι εμείς ε, για ένα αποτέλεσμα. Ο Πέτρ Γκέζεκ. Ευχαριστώ. Για να συμπληρώσω, θα όσο είπε ο ένα από τα βασικά συμπεράσματα από αυτό το έργο είναι ότι πολλές από τις πρακτικές στα Panama Papers δεν θα είχαν συμβεί καθόλου ή θα είχαν συμβεί σε πολύ μικρότερο βαθμό εάν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν αναλάβει τις ευθύνες τους με τρόπο πιο ενεργό αν είχαν λάβει περισσότερες πρωτοβουλίε και αν είχαν εφαρμόσει στην πράξη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θεωρούμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης, το γράφουμε στην έκθεση ούτως ή άλλως, στις περιγράφους 57 και 58 που αναφέρονται στην εφαρμογή της ε, οδηγίας 3 περί ξεπλήματος. Αν και προωθήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις στα κράτη-μέλη, δυστυχώς διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις ή ελλείψεις στην εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης, η ποιότητα ή αν θέλετε η αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασίας υπερβάση είναι αμφιβολή σε πολλέ χώρε. Πολλέ χώρε λοιπόν δεν εφάρμοσαν την οδηγία ε, AMLD 3, κάτι το οποίο κρατείνει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή με την σειρά τη δεν φρόντισε την ομαλή μεταφορά και εφαρμογή. Στην παράγραφο 5 παρατηρούμε ότι οι εθνικές αρχές δεν επέβλεψαν αποτελεσματικώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πριν την αποκάλυψη των Panama και μάλιστα δεν επέβαλαν επαρκείς κυρώσεις επί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είχαν ε, διαπιστωθεί να παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία αλλά και την οδηγία. Παράγραφος 135, εκεί συμπεραίνουμε ότι η απουσία συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, τουλάχιστον, αποτέλεσε εμπόδιο. το θεωρείται παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας, καθώς εν τέλει η έλλειψη συνεργασίας ήταν εμπόδιο στην ερευνά μας. Εξού σημαντικό και ίσως πιο ανησυχητικό θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφιερώνει, δεν πάνε αρκετούς πόρους για να διεκπαιρεώσει τον ρόλο της, του επόπτη δηλαδή και για την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη. Όπως είδαμε και με την κατεξοδότηση πράξη για τις τρίτες χώρες. Εκεί έχουμε περίπτωση κακοδιοίκησης. Και επίσης φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντελεί τέλει το έλεγε αυτό υπόψη τη και προετοιμάζει τις μελλοντικέ τη ενεργείες. Όσον αφορά τι συστάσεις μας, χαίρομαι ότι ευκολώς συμφωνήσαμε επί συγκεκριμένων συστάσεων με τον συνάδελφο, με τον Γέπε. Η συστάσει είναι βασικά περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη ρύθμιση των αγορών, περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους. Στην έκθεση λοιπόν με την λύπη μας για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν βοήθησε να αποκαλύψουμε τους πραγματικούς δικαιούχους των καταπιστευμάτων, ούτε ενδιαμέσους που διευκολύνουν την φοροποφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Χρειάζεται λοιπόν επίση καλύτερη ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών με συγχωρείτε, μεταξύ φορολογικών αρχών αλλά και μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Χρειάζεται περισσότερε προσπάθειε σε επίπεδο φορολογική διοίκηση, ε, αλλά και ακόμη περισσότερο, όπω ε, προείπα, στι ε, μονάδε συγκέντρωση πληροφοριών για τα χρηματοοικονομικά. Όσον αφορά του καταγγέλλοντε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή, πραγματικά ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του όσον αφορά την διαθεσμική συνεργασία και τα δικαιώματα των ε, διερευνητικών επιτροπών, πιστεύω ότι η Επιτροπή μας χρειάζεται σοβαρές αλλαγές για να γίνει πιο αποτελεσματική στο μέλλον. Οι κυβερνήσεις πρέπει να τον δουν λίγο πιο σοβαρά και δηλαδή είναι το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα καλό παράδειγμα. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις, να υπενθυμίσω ότι μερικές μπορούν να υλοποιηθούν αμέσως βάσει των συστάσεων της οδηγίας, της AMLD. Άλλες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του τριμερούς διαλόγου. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνουμε ότι κάποια τουλάχιστον κατημέλη θα δουν εμπόδια στην εφαρμογή περισσότερη διαφάνειας. Ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες θα καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της έκθεσης και ότι αυτό θα ενισχύσει την εντολή μας για την αναθεώρηση δηλαδή και εν ώψη των συνομιλιών για την αναθεώρηση της οδηγίας. Θεωρώ ότι η ικανή πολιτική υποστήριξη θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε όλα αυτά στην πράξη. Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η έκθεση είναι η καλύτερη που έχουμε βγάλει ποτέ και ζητώ σχετικώ την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές για τις παρουσιάσεις τους. Και θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εμεί ε, από την Επιτροπή μας μπορούμε να διατυπώσουμε τροπολογίε ε, ή συστάσει και για τα δύο τμήματα τη ε, δουλειά σα. Στην Ολομέλεια μόνο στι συστάσει μπορούν να γίνουν συμπληρώσει. Θέλω να το τονίσω αυτό. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ μέσα στην Επιτροπή μέλη μπορούν να, να διατυπώσουν τις προτάσεις τους και τις τροπολογίες τους για κάθε κομμάτι των εγγράφων σας, ενώ στην Ολομέλεια μόνο στις συστάσεις. Ο κύριος ε, Νίτερμαϊρ είναι εδώ τώρα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως και ηγητής. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ξεκινώντας θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για μια δουλειά μακροχρόνια, σκληρή, σε ένα πολύ δύσκολο θέμα που εντάσσεται και στις ε, συνεχιζόμενες προσπάθειές μας ε, για την βελτίωση του θεματολογίου του σχετικού με τη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώ λοιπόν με την έκθεση, η οποία νομίζω καλύπτει επί της ουσίας όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τα έγγραφα του Παναμά, αλλά και θέματα νομοθεσίας των τελευταίων ετών, νομοθεσίας που εισήχθη για να καλυφθούν κάποια κενά νομοθετικά. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις και αποστολές στο πλαίσιο της Επιτροπής μας, που και αυτές αντικατοπτρίζονται εδώ. Το υλικό το οποίο μας διατέθηκε ήταν τεράστιο. Οι συνεισηγητές μπόρεσαν με πολύ μεγάλη επιδεξιότητα και τα πορίσματά τους και τις διαπιστώσεις να τις καταγράψουμε σας στις εκθέσεις. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω για τη βούληση να συμπεριλάβουν ε, μετά τη συνεδρίαση των σκιωδών συγητών τα αιτήματά μας που διατυπώθηκαν αμέσω μετά τη δημοσίευση της έκθεσης. Κάποια στοιχεία πιστεύω θα μπορούσαν να ε, διαμορφωθούν κατά καλύτερο ή σαφέστερο τρόπο και πάνω απ' όλα το θέμα του χρονικό μας ενδιαφέρει. Έχουμε να κάνουμε με ένα ε, όγκο εγγράφων, στην περίπτωση των ε, εγγράφων του Παναμά, που ανάγονται μέχρι και το 1970. του 70. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι πιο σαφής η παρουσίασή τους και τα πορίσματα να ανάγονται επίσης την ίδια χρονική περίοδο. Δεν μπορεί όλα τα έγγραφα να έχουν την ίδια σημασία, αν έχουν ήδη καλυφθεί παραδείγματι από την εντωμεταξύ ε, εισαχθής αναμοθεσία. Δεν πρέπει να συζητούμε τώρα υποθέσει που ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν. Ε, ο χρονικό λοιπόν παράγων θα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο να καταλήξουμε και στα θεμητά και αιτιολογημένα συμπεράσματα και πορίσματα. Και για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις μάλλον που διατυπώνονται θα τις κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για να διατυπώσουμε τις τροπολογίες μας. Αλλά δεδομένου ότι είναι τόσο περίπλοκο όλο αυτό το θέμα και πολλές οι ε, πληροφορίες θα πρέπει να διαβάσουμε πιο προσεκτικά για τις συστάσεις λοιπόν που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μόλις έχουν κέρια σημασία πιστεύω για τη δουλειά μας και στις επιτροπές τάξη 1 και τάξη 2, άλλωστε το διατυπώσαμε μέσα από, τα, από τις συστάσεις μας. Είναι αιτιολογημένες πολλές από αυτές τις συστάσεις, ε, ωστόσο ε, έχουν διατυπώσει και προτάσει για νομοθετικέ τροποποιήσεις, οι οποίε θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. στι συστάσεις, στις προτάσεις συστάσεων, οι δύο συνεισηγητέ έχουν επιτύχει τη σύνδεση με την κύρια έκθεση και την ε, παραπομπή σε κάθε περίπτωση ποια σύσταση αναφέρεται σε ποιο σημείο της έκθεσης. Όσον αφορά τις συστάσεις, συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές, ιδιαίτερως εκεί όπου γίνεται λόγος για περισσότερη προσοχή σε θέματα που έχουν να κάνουν με αυτούς που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, αλλά και την διερεύνηση της ισχύουσας νομοθεσίας ε, όπως αυτή έχει εισαχθεί στα κράτη-μέλη. Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι το σημείο 5 του κανονισμού που έχει ήδη περάσει τριμερή διάλογο να υπογραμμιστεί, να ενισχυθεί και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εργαστεί έτσι ώστε να καταλήξει σε συμβαστική λύση με το Συμβούλιο γιατί ο κανονισμός αυτός μπορεί να κλείσει πολλά παραθυράκια που έχουν εντοπιστεί στην νομοθεσία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει απολύτως σεβαστή η εντολή της Επιτροπής ΠΑΝΑ, δηλαδή να μην υπερβούμε το πλαίσιο της εντολής αυτής, αλλά και να καλύψουμε όλα τα θέματα τα οποία έχουν αναφορά μόνο στην δική μας Επιτροπή και όχι σε εργασίες άλλων φορέων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των συστάσεων ε, και συγκεκριμένα να απευθυνθούν αυτές οι συστάσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να ληφθούν από αυτά τα όργανα ε, σοβαρά υπόψη για να αναλυφθεί η απαιτούμενη δράση. Βεβαίως στις συστάσεις κάποια σημεία δεν με βρίσκουν όπως σύμφωνο ή θα χρειαζόταν ε, για να τα δεχθώ περισσότερο διάλογο. Θα τα καλύψουμε στις τροπολογίες μας. Επί παραδείγματι δεν ξέρω αν είναι ευχερής η εγκαθίδρυση νομοθεσίας για το τι συνιστά ανήθικη δράση. Επίσης ε, στην εισαγωγή της Ευρωπαϊκής ΦΑΤΚΑ που ζητούν οι συνεισηγητές ή της εξωτερικής ανάθεσης της αρχής της ε, πρόληψης δεν ξέρω πόσο καλά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Απαραίτητο είναι πάντως η αρχή της πρόληψης να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ικανοποιητικά. Πολύ ευχαριστώ όμως να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα που με απασχολούν. Δεν συμφωνώ απαραίτητα ότι θα πρέπει να περάσει κάθε λύση μέσα από νομοθετική παρέμβαση. Νομίζω ότι και η αυτορύθμιση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και μπορούμε χάρη σε αυτήν να περιοριστούμε στην ε, εισαγωγή μόνο θεμά, στην, ε, στην ομοθεσία μόνο θεμάτων που έχουν ε, καθαρά νομοθετικό χαρακτήρα και τα υπόλοιπα να περάσουν στην αυτορύθμιση. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ιδιαίτερως ευχαριστώ όλη την Επιτροπή, τον Πρόεδρο, τη Γραμματεία για την πολύ σκληρή δουλειά, αλλά και όλους τους συναδέλφους με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στην εξαίρετη δουλειά των δύο συνεισηγητών. Η δουλειά αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή βάση για την ε, περαιτέρω έκθεση που θα υποβάλουμε στην ε, Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ Λούντεκ, λέει ο Πρόεδρος. Όσον αφορά την εντολή, είναι σχετικά ευρία η διατύπωσή της γιατί έχουμε και την συνέχιση των εργασιών ε, των Επιτροπών Τάξε 1 και 2 στην αυτορύθμιση από τις διερευνητικές αποστελές και κυρίως αυτή του Λουξεμβούργου αποδεικνύεται ότι από 300 ε, δικηγόρους μόνο μία περίπτωση επαληθεύθηκε, ελέγχθηκε. Εν πάση περιπτώσει όμως χρήσιμο το σχόλιο σου. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση και θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση συνεργασίας. Εκ μέρους της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Σαμπάτσκι δεν είναι εδώ παρόν, ούτε και έχει ε, ορίσει εκπρόσωπο ε, για να τον αντιπροσωπεύσει. Φαντάζομαι ότι είναι στο δρόμο επιστρέφοντας από την Κύπρο. Ο Κρέσπο παρακαλώ. Πού είναι, να το περάστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρώτα πρώτα ευχαριστούμε τους εισηγητές, διότι μας παρουσίασαν αυτό το έγγραφο το οποίο νομίζουμε αποτελεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή του θέματος και είναι αξιόλογες οι Προτάσει, Πρώτα απ' αυτά ο κόσμο. παραμένει, περιμένει πολύ περισσότερα από εμά. Έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα όσον αφορά την χρησιμότητα του Κοινοβουλίου ιδίω μετά από όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Και θα ήθελα να σα θυμίσω και έλεγε ο Βίκτορ Ογκό. Έχει πολλά ονόματα το μέλλον για του ε, αδυναμου, είναι κάτι το άπιαστο για του τολμηρού, είναι κάτι το άγνωστο και για του ε, θαραλέου είναι μια ευκαιρία. Σήμερα, συνάδελφοι, θα πρέπει όλοι να επιδείξουμε θάρρος. Νομίζω ότι ε, αυτό το έγγραφο μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με τη διαδρομή που έχουμε χαράξει και επομένω θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία αναφέρονται και εκκρεμούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προχωρήσουμε. Και θεωρούμε ότι το εξέλιγμα χρήματο και οι φορολογικέ απάτε είναι οικονομικός οικονομική τρομοκρατία. Γιατί αυτό κάνουν, χρηματοδοτούν ε, εγκληματική δράση και, και επίσης ε, υπονομεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα και την φορολογική βάση. Οπότε θα πρέπει αυτό να γίνει η Ευρωπαϊκή να έχει ένα τέτοιο πλαίσιο για να ελέγχει την κίνηση κεφαλαίων, τους διάφορες ωραίες των κεφαλαίων και να υπάρχει ε, μόνιμη, ε, ε μόνιμος φορολογικός και θα πρέπει επίσης να ε, μπορέσουν να έχουμε ανταλλαγή των παρικών μοντέλων σύμφωνα με τις ανάγκες της ε, πλειοψηφίας του πλανήτη. Είναι απαράδεκτο να ανεχόμαστε ε, αυτού του είδους τα φορολογικά κενά από κάποιες ε, χώρες και θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει φορολογικό ντάμπινγκ. Όλοι οι εγκληματίες από τη χώρα μου στέλνουν τα χρήματα στην Αντόρα και στην Ελβετία και αυτό δεν γίνεται τυχαία γιατί αυτές οι χώρες και άλλες δεν συνεργάζονται για τα φορολογικά όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν ε, κάποιοι συντελεστές οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί και υπάρχουν τρόποι ε, ούτω ώστε να αποκρύπτουν τους ε, πραγματικούς δικαιούχους και έχουν ως πρόφαση το, το, το απόρριτο, το επαγγελματικό απόρριτο, αλλά δεν ασκείται κάποιο είδους δέουσα επιμέλεια για αυτό που πρέπει να κάνουν. Άρα θα πρέπει να αναστείλουμε προσωρινά τις σχέσεις με αυτές τις χώρες. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της διαδικασίας, της διαδικασίας χωροποφυγής και πλησίματος του χρήματος. Θα πρέπει επίσης το μέγεθος των ποσών να καθορίσει ε, την ευθύνη και όχι ο αριθμός των εταιριών που εμπλέκονται. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος και για αυτό και για τις φορολογικές και ποινικέ ευθύνε να έχουμε ένα διεθνές μητρό των πραγματικών δικαιούχων. Να ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις από την τάξη 1 και την τάξη 2, επίσης η αναθεώρηση της τέταρτης οδηγίας κατά του ξεπλήματος θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα όσα προτείνουν οι ειδικοί στις ακροάσεις μας οι οποίοι έλεγαν θα πρέπει να έχουμε ως κυρώσεις την ε, αναστολή λειτουργίας τραπεζών τους της άδειας λειτουργίας τράπεζας και που γνωρίζετε όλη η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη θα πρέπει τους ε, ενδιάμεσους και τους ε, διευκολύνοντες έτσι να τους ονομάζουμε και όχι ε, μεσίτες και όχι μεσάζοντες. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει με βάση την ε, λίστα που υπάρχει, τη λίστα γκάφη, να δούμε τι γίνεται με τις χώρες που έχουν συντελεστές κάτω από συγκεκριμένο κατόφλι και επίσης θα δούμε τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Και πάλι ευχαριστούμε για αυτό το πλαίσιο εργασίας που προτείνεται και με κάποιες τροπολογίες πιστεύουμε θα ενταχθούν και αυτές στο κείμενο που νομίζω ότι θα είναι ένα λιθαράκι για να θεσπιστεί νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε αυτά τα σημαντικά φαινόμενα. Και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα δείγμα θάρρους προς τον κόσμο που προσβλέπει στη δράση μας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφα. Εκ μέρους της ΓΚΟΑ. Σε ένα σημείο θα ήθελα να σε διορθώσω ότι οι φορολογικοί συντελεστές εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι φορολογικό δίκαιο δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε ή τουλάχιστον δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει ε, γιατί υπάρχουν πολλές αντιστάσεις αλλά πάντως πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη φορολογική βάση και συντελεστές ε. Εάν, επί παραδείγματι, η Μάλτα μειώνει κατά 30% το φορολογικό της συντελεστή για τους αλλοδαπούς, δεν νομίζω ότι προσφέρει ε, ισότιμες φορολογικές συνθήκες. Αν θες να απαντήσεις. Το ξέρω, Πρόεδρε. Αλλά δεν είπα ότι θα, κάνουμε, θα νομοθετήσουμε, αλλά να δώσουμε επιχειρήματα στις χώρες, στο Συμβούλιο, σε όλε όργανα, ούτω ώστε τελικά να καταλήξουμε να μπορούμε να νομοθετούμε. Γι' αυτό είναι το σημαντικό. Πρόεδρο. Εντάξει. Η κυρία Μόλι Σκοτ Κάτω, εκ μέρου των Πρασίνων, παρακαλώ. Θα συμφωνήσω με του προλήθεντε. Είναι πολύ και σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη συνεργασία της. ω προ την διαδικασία τώρα. Υποστηρίζουμε να εκδοθούν τρία κείμενα για το έργο μα για τα ευρήματα και για τις συστάσεις. Υπάρχει μια σχετική επικάλυψη βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή βάση όλα αυτά να προχωρήσουμε. Η επισκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκθέσεις μας, ε, αλλά να σκεφτούμε και αυτούς που θα διαβάσουν όλα αυτά σε μερικούς μήνες και όχι μόνο εβδομάδες. Το θέμα είναι να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κρίνουν το έργο μας. Ως προς το περιεχόμενο, συμφωνούμε με τα βασικά συμπεράσματα όσον αφορά φοροδιαφυγή, φοροποφυγή, διαμέσους, ξέπλυμα και ούτω καθεξής. Εν γέννη, συμφωνούμε και με το συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειψη επαρκού ικανού νομοθετικού πλαισίου αλλά και εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και ότι απαιτείται περαιτέρω εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει επίση τα κράτη-μέλη να το πάρουν απόφαση να συνεργαστούν με την Επιτροπή Πάνα. Αν και οι τα συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει παράβαση της οδηγίας ή της οδηγίας για το ξέπλυμα, θεωρούμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις κακοδιοίκηση και αυτό το συμπέρασμα το ξαναβλέπουμε με τους δικηγόρου μα και θα σα ενημερώσουμε για το πού θα καταλήξουμε. Ορισμένοι πιστεύουν ότι υπήρξε παράβαση των κανόνων τη τρίτη οδηγία για το ξέπλυμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα υποβάλουμε σχετικώ τροπολογίε. Λείπει επίση ε, συγκεκριμένη αναφορά στην κακοδίκηση από τα κρατημέλη. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους αναφέρουμε χώρε με το όνομά του. Ας πούμε, η ομάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρηση της Μάλτας μα λέει ότι η αστυνομία δεν κινήσε όλες τις υποθέσεις. Επίσης, όσον αφορά την τέταρτη οδηγία στην Γερμανία και εκεί οι πρακτικές παραβαίνουν τους κανονές σε ανώτερο επίπεδο. Με αντικείμενο τους ε, Όσον αφορά τις ε, συστάσεις και προτάσεις, θα υποβάλουμε ορισμένες τροπολογίες σε αυτό που θεωρούμε γενή κοινή βάση. Πρόκειται για την ενίσχυση των ε, ικανοτήτων μας έρευνας. Το Συμβούλιο, το ξέρουμε, στην αρχή ήταν διστακτικό στο να συνεργαστεί με την ΠΑΝΑ. Δεν ήθελα να περάσουν στα χέρια μας αρμοδιότητες, γι' αυτό προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες μας με άλλους τρόπους. Οι συστάσεις μας επίσης αναφέρονται στα βασικά ζητήματα των Panama Papers. Το θέμα είναι πώς ε, αξιοποιούνται από διάφορου τα ευρωπαϊκά κρατημέλη και δει το ΣΥΡΙΠ του Λονδίνου που είναι εγκαταστημένη μισή χρηματοπιστωτική φορείς. Πρέπει ο τομέας αυτός, ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών να τεθεί εν γέννη στην υπηρεσία όλου του πλανήτη. Επίσης, περιμένουμε ενεργητική δράση από τους ενδιαμέσους. Αυτό δεν αναφέρεται εδώ. Θα ήθελα λοιπόν πιο συγκεκριμένες προτάσεις στον τομέα αλλά και στη γενικότερη προσέγγιση που αφορά τη γνώση όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά το λεγόμενο tax planning, τον ε, φορολογικό σχεδιασμό κλπ. Δεν έχω χρόνο, το καταλαβαίνω, αλλά μισό λεπτό πρόεδρε, ένα λεπτό. Να είμαστε ενωμένοι. Δεν είμαστε εδώ για να υπεραμεινθούμε εθνικών συμφερόντων. Δουλεύουμε για όλου του Ευρωπαίου. Πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ είμαι Βρετανίδα, όπω γνωρίζετε, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που βρήκαμε στα Panama Papers είναι ισχυρέ ενδείξει ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στη σχέση μεταξύ του Λονδίνου και των διαφόρων χρηματοπιστωτικών αγορών. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όλα αυτά βεβαίω πρέπει να συμφωνηθούν πριν το Brexit. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε με την σύσταση αυτή, ειδικά. Αυτά προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συζητήσει με εσά και με του Κιώδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συναδελφέ Ήθελα να τονίσω το τελευταίο αυτό σημείο που αναφέρατε, γιατί το έχουμε ακούσει και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι παντού ισχύουν οι κανόνες, αλλά οι εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ελέγχουν την επικράτειά του ολόκληρο. Ο κύριος η FTT. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τους δύο συγκητές. Έκαναν και αυτή τη φορά εξαιρετική δουλειά προάγοντας τον αγώνα μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιρετικές συστάσεις τους. Ίσως θα έπρεπε να διατυπωθεί ακόμη μια σύσταση. Να γίνονται σεβαστές οι συστάσεις, δηλαδή του Κοινοβουλίου την ώρα που διατυπώνεται η νομοθεσία. Γιατί και στην προηγούμενη ολομέλεια το Κοινοβούλιο έδωσε το στίγμα της, ε, με τις προτάσεις για τη φορολογία. Και νομίζω ότι αυτό που συνέβη ήταν ένα βήμα οπισθοδρόμησης υπέρ των πολυεθνικών. Ένα συνταρακτικό βήμα οπισθοδρόμησης. Έτσι λοιπόν το να κάνουμε τόσες προσπάθειες, τάξε 1, τάξε 2, πάνα και μετά να βρισκόμαστε να λαμβάνουμε αποφάσεις με τον λανθασμένο τρόπο, νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γι' αυτό θα ήταν καλό να ε, εισαχθεί στις συστάσεις μια διαδικασία απολογισμού ή λογοδοσίας αναχώρα, μια επαλήθευση, εν πάση περιπτώσει, φιλόδοξη για το αν τήρονται αυτές οι συστάσεις. Όπως άλλωστε προτάθηκε και στην Ολομέλεια σε κάποια ψηφοφορία. Για την μαύρη λίστα, για την άρση της ισοδυναμίας με τις χώρες αυτές, τρίτες χώρες. Ίσως θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο αυστηροί, θα διατυπώσουμε τις σχετικές προτάσεις για τον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Μας φαίνεται πολύ παράξενο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικό της κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνει καμία από τις χώρες που έχουμε εμείς εξετάσει στην Επιτροπή μας και στα έγγραφά μας. Πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί. Επίσης, ένας καταλόγος φορολογικών παραδείσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί λοιπόν. Όπου έχουμε εμείς άμεση αρμοδιότητα, δεδομένου ότι υπάρχει και εσωτερική στρέβλωση του φορολογικού ανταγωνισμού και βέβαια οι καταστροφικές συνέπειες κοινωνικές και οικονομικές που προξενούν αυτές οι στρεβλώσεις. Συμφωνούμε επίσης ως προς την προσέγγιση τη σχετική με τις τράπεζες ή τους μεσάζοντες που μπορεί να έχουν ε, να επιδείξουν, μη, ε, να μην, επιδείξουν ε, απουσία διάθεση συνεργασίας με συνέπειες που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και στην ανάκληση της άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών. Οι τράπεζες είναι μεταξύ εκείνων που ωφελούνται τα μάλλα από αυτά τα προβλήματα, από αυτά τα σκάνδαλα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού αυτές διακινούν το χρήμα, θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί απέναντί τους. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ισχυρό το λόμπι των τραπεζών βεβαίω, αλλά καθήκον μα, καθήκον των πολιτικών, είναι να βρούμε λύσεις σκληρές και αποφασιστικές. Στην ενίσχυση της ε, νομοθεσίας για την καταπολέμηση της ανακύκλωσης εσόδων από παρανόμες δραστηριότητες και εδώ πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις σχετικές πληροφορίες ε, με διάκριση μεταξύ των ε, κερδοσκοπικών και μη ε, ενώσεων ή οργανώσεων ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Πάνα, ε, στην ε, επίτευξη του έργου μας. Όπως είπε και η συνάδελφος Μόλι, θα πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ αυστηρό τρόπο τους λόγους και να τους καταγράψουμε σε ένα έγγραφο. Και τελευταίο, για τον κώδικα συμπεριφορά θα ήταν σκόπιμο στην έκθεση να συμπεριληφθεί και μια πρόταση για μια εις ανάλυση των 19 ε, ετών εργασιών που μας απασχόλησαν με μία πρόταση που θα οδηγήσει και σε ριζική αναθεώρηση του κώδικα συμπεριφοράς ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι όπως περιγράφονται. Ασφαλώς και όλοι συμμερίζονται το έγγραφο στις γενικές του γραμμές. Ασφαλώς και ο καθένας θα μπορούσε να προσθέσει ένα συγκεκριμένο σημείο ή μία παρατήρηση. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το Κοινοβούλιο αλλά και τα θεσμικά όργανα γενικά όταν έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή να μην... Ε, επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, αλλά να προχωρούν με τρόπο θαραλέο, σε σχέση με αυτά που είδαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ας ενθαρρύνουμε αυτούς που θέλουν να εργάζονται με τρόπο σοβαρό με τις εκθέσεις αυτές. Ακριβώς αυτή θα ήταν μια πρόσθετη σύσταση. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα υπάρξει μια τέτοια ευκαιρία, ας μην πάει χαμένη. Γιατί διαφορετικά ε, χάνουμε την ευκαιρία για, τον, ε, για την άσκηση από πλευρά του Κοινοβουλίου των Θεσμικών Οργάνων του Ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάλη, λέει ο Πρόεδρος, ε, σε σχέση με τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των φορολογικών παραδείσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θυμούμε καλά, ότι είχε πει πως φορολογική παράδοση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνονται μόνο στον κατάλογο αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να το δεχθούμε. Η κυρία Κάπλ, η e ΕΝΕΦ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ θερμά τους δύο συνεισηγητέ για τις προτάσεις τους. Είναι πληρέστατες έχουν ε, καλή ισορροπία, δίνουν έμφαση στα κατάλληλα, στα σωστά σημεία και με την αποστολή που είχαμε τώρα στην Κύπρο, άλλωστε το, ξανα, το ξαναείδαμε, με μεγάλη αδημονία βλέπουμε ότι περιμένουν όλοι το είδαμε και στην Κύπρο συγκεκριμένα και τα κράτη-μέλη αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, παραδείγμα η Financial Intelligence Unit, FIU, περιμένει με αδημονία να δει τι θα φέρει αυτή η έκθεση, της, πώς συγκεκριμένα θα διατυπωθεί και όταν θα είναι έτοιμη η έκθεση δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και για τους εμπλεκόμενους φορείς, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο κάνουμε δουλειά γιατί ακριβώς αυτό το θέμα της καταπολέμηση της φοροαποφυγής και κάθε συναφού ζητήματος των ζητημάτων δηλαδή που προέκυψαν ε, και με το σκάνδαλο του Παναμάλα και με τα υπόλοιπα ε, μας ε, υποχρεώνουν να επιτελέσουμε στον ύψιστο δυνατό βαθμό το έργο μας. Είναι πολλές οι προσδοκίες, πρέπει σε αυτές να ανταποκριθούμε και έτσι στα συμπεράσματα ε, επισημάνονται κάποια, επισημαίνονται κάποια σημεία τα οποία μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν με την τάξη αλλά και στο σκάνδαλο του Πανωμά ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία πολύ περισσότερο και μεταξύ των κρατών μελών χρειάζεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ακόμη και με την ε, ε, επαπειλή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν ε, συνεργάζεται κάποιο ε, αρχή και αυτό νομίζω και η ομάδα εργασίας για τον κώδικα συμπεριφοράς θα πρέπει να το λάβει υπόψη, να να αναφέρετε και στα συμπεράσματά σας γιατί στο παρελθόν είχαμε επισημάνει και δει αδυναμίες που ελπίζουμε ότι με τη νέα ηγεσία στην ομάδα εργασίας για τον κώδικα συμπεριφοράς θα ξεπεραστούν. Επίσης, ε, κάτι ακόμη που θα ήθελα να επισημάνω για την τελική έκδοση της έκθεσης, σε πιο συγκεκριμένου όρους λίγο πολύ, γιατί δεν είναι πάρα πολύ σαφές για μένα το τι προβλέπεται σε σχέση με το μαύρη λίστα. Ε, είχε πει η Επίτροπος Γιώροβα ότι θα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κατάλογοι. Ο ένας θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίας και άλλο ένας που θα καλύπτεται από την οδηγία για τα τρίτα κράτη που εμπλέκονται σε νομοποίηση ε, προϊόντων εγκλήματος, παράνομων εσόδων. Ε, νομίζω ότι και σε συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές μπορούμε να ε, καταρτήσουμε τους καταλόγους αυτούς. Δεν χρειάζεται να μείνουν ε, οι καταλόγοι αυτοί μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε και με την, στην Επίτροπο το επισημάναμε αυτό και νομίζω το αντελήφθη για τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο, την Ευρωπαϊκή Μαύρη Λίστα θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι το σκόπιμο ή αν είναι καλύτερο να πούμε ότι τα κράτη τα οποία δεν συνεργάζονται είναι κράτη τα οποία ε, θα πρέπει να προσβληθούν με την διαδικασία επί παραβάση να προσταθούν δηλαδή ενώπιον του δικαστηρίου με την ε, διαδικασία παραβάση, αν δεν αλλάζουν στάση. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει το σημείο στο οποίο κατακρίνονται οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, όπου δεν διαθέτουν ε, επαρκές προσωπικό ή άλλους πόρους για την δίωξη των σχετικών αδικημάτων ή ε, προβλημάτων. Θα πρέπει δηλαδή να τονίσουμε το γεγονός ότι η απουσία, η έλλειψη, η αδυναμία σε πόρους μπορεί να επιδεινώσει ακόμη το πρόβλημα και γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθούμε στις εθνικές αρχές που θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη αυτή. Στο δε σημείο 25, Λουξεμβούργο, Κύπρος και Ηνωμένε Πολιτείε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό γιατί από τις διερευνητικές αποστολές που κάναμε ε, στις χώρες αυτές μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι δεν ε, είναι ε, αμεληταία τα προβλήματα και πρέπει να εξετάσουμε μεγάλη προσοχή τι συμβαίνει στις χώρες αυτές για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάλι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλογος ε, εκείνων που δεν τηρούν τους κανόνες, μαύρη λίστα δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η FIU και σε συνεργασία με τη Europol, γιατί το είδαμε και στην Κύπρο πάλι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας Edmond. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί και άλλο ένα σημείο σε σχέση με τους μεσάζοντες. Στο 113 συγκεκριμένα σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταπιστεύματα μπορούν να είναι σημαντικοί ε, μεσάζοντες και θα πρέπει και σε αυτά να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Ε, το λεγόμενο σκιώδες τραπεζικό σύστημα θα πρέπει και αυτό να υπαχθεί σε πιο αυστηρούς κανόνες για να εξασφαλιστεί μέχρι στη δυνατή διαφάνεια. Επίσης, το είπα ήδη, θα το επαναλάβω, ε, καλύπτονται στο κείμενο τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε δει στο παρελθόν και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για να δώσουμε και τα σχετικά κίνητρα στα κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη συνεργασιμότητα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Έτσι εξαντλήσαμε τον κατάλογο των εδώ παρόντων σκιωδών εισηγητών, γιατί ο κύριος Σαμπάτσκι ακόμη δεν έχει έρθει. Και έτσι περνώ στους ομιλητές εκ μέρου των ομάδων τους, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού ε, κόμματος, ο κύριος Φαντέν Κελάρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, φέρω εκτός τον θαυμασμό μου για το δυναμισμό των ε, συνεισηγητών. Είναι πλήρες το κείμενό τους, πρόκειται να αποτελέσει εξαιρετική αφετηρία για τις εργασίες μας. σύμφωνα με τον κύριο Νίντερ Μάγερ θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα, θα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε το κείμενο, να έχουμε συγκεκριμένη διατύπωση στην έκθεση να αποτελέσει κάτι πιο αποτελεσματικό επικοινωνιακά. Τώρα, όσον αφορά τους ε, ενδιάμεσους, τους διαχειριστές περιουσιών, σε σχέση με τις κυρώσεις συμφωνώ με όσα άκουσα, δεν θα προσθέσω τίποτα σήμερα. Τώρα, τρία δευτερεύοντα σημεία, ε, τα οποία έχω επισημάνει, σε μια πρώτη νόηση του κείμενου πρώτα-πρώτα, το νομοθετικό πλαίσιο για το ξελίγμα χρήματος θα πρέπει πάνω απ' όλα να φροντίσουμε να υπάρχει αποτελεσματική και λογική εφαρμογή του νόμου. Λέει proper implementation το κείμενο Νομίζω ότι χρειάζεται κάτι συνεκτικό, κάτι λογικό, κάτι συνεπές. Είναι θέμα συνέπειας και όχι μόνο ορθότητα, ας το πούμε έτσι. Ας πούμε consistent, αν ήταν στα αγγλικά. Και αν υπάρχουν ορισμοί, αυτοί να είναι ταυτόσιμοι σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, όσον αφορά αυτή την ε, μονάδα, αυτή την ε, υπηρεσία πληροφόρων για τα χρηματοοικονομικά, την FIU. Φιλόδοξη αυτή η πρόταση, αλλά προσοχή γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα. Οπότε θα πρέπει να τονίσουμε το ότι θα πρέπει να επιστατευτούν περισσότεροι πόροι για τέτοιες financial intelligence units σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών. Ε, επίσης, να δούμε τι θα γίνει με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις οδηγίες DAC. Θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά. Και επίση οι εθνικές αρχές χρειάζονται κάποιους πόρους για να γίνει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτές τις τρεις ε, παρατηρήσεις είχα. Θα παρακολουθήσω τις εργασίες μας και εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους συγκεκριμένους και τους σκιώδες. Ευχαριστώ. Η Έλλη Σλάιν τώρα, εκ μέρου Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Είναι στον κατάλογό μου. Ας περιοριστούμε λίγο πολύ στι δίλεπτε παρεμβάσεις, παρακαλώ. Ε, μικρό. Ευχαριστώ πολύ τον Γέπε. Χαίρομαι ότι θίξαμε και την διεθνή διάσταση καθώς και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές είναι που πλήττονται κατά κύριο λόγο από την φοροποφύγη και φοροδιαφυγή. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ενιαία διεθνή λύση. Όπω είπαν και οι συνάδελφοι, οι κανόνε είναι αποτελεσματικοί όταν είναι ενιαίοι, όταν έχουμε κανόνες χωρίς εξαιρέσει, όπως κάνουμε στο παρελθόν. Πρέπει την διαδικασία αυτή να θέσουμε υπό έναν φορέα των Ηνωμένων Εθνών. Οι κανόνε του ΩΣΑ, ξέρετε, δεσμεύουν μόνο τις χώρες μέλη του ΟΣΑ. Όμως δεν ασκούμε και καμιά πίεση στις χώρες του ΟΣΑ όταν δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν με το πρόσημο πολλές φορές ότι δεν έχουν προσωπικό ή χρήματα για να συμμορφωθούν. Πολλές φορές αυτό είναι αλήθεια, ακόμα και για ανεπτυγμένες χώρες. Δείτε την κοινή έκθεση του ΟΣΑ για τα κοινά πρότυπα, τους κοινωνικούς, τους κοινούς κανόνες εδώ υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να συλλέξουν καν τα στοιχεία. Χρειάζεται τεχνογνωσία, χρόνος, κόπος για να φτάσει κανείς στα επιθυμητά επίπεδα όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Έτσι όπως ε, ζητάει το Κοινοβουλίο στην έκθεση της 15ης Ιουλίου. Έχουμε και κατάλογο με τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες. Εκεί μην ξεχνάτε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν φτωχές χώρες όπως η Λιβερία αλλά και κάποιες πολιτείες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην νομίζετε. Είναι εύκολο να θεσπίσει νέες υποχρεώσεις. Και εν πάση περιπτώσει μετά μπορούμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά αν και πώς χρησιμοποιούνται οι σχετικές συνθήκες, περιφορολογίες κλπ. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αναπτυσσόμενες χώρες χάνουν εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ακυρώνεται η δική μας αναπτυξιακή πολιτική. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας. Επόμενος. Λέωνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ε, συνεισηγητές για, το, για την εξαντλητική αντιμετώπιση και διερεύνηση του θέματος. Νομίζω συνοψίζουν ε, με βέλτιστο τρόπο τη συζήτηση μας εδώ. Δύο πράγματα πάντως, με την ευκαιρία. Στο 2-4 έχουμε κατάλογο χωρών ή είναι στο 2-2, δεν θυμάμαι. Θέλει λίγο δουλειά αυτός ο κατάλογος. Να πάμε και στο 2-1. Χρειάζεται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στο, στο επίπεδο των, της ΦΑΤΦ. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη σύγκριση μεταξύ, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στο απειρόβλητο αυτούς τους γνωστούς φορολογικούς παραδείσους επίσης να δούμε με ποιους τρόπους θα συνεχίσουμε το έργο μας στο μέλλον. Τι είδου πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε τα επόμενα ας πούμε πέντε χρόνια. Δεν έχω τις απαντήσεις, έτσι, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Εάν το αφήσουμε το όλο πράγμα θα χάσουμε την ορμή, θα κυρώσουμε το έργο μας και να μην ξεχνούμε και τους καταγγέλλοντες δημοσιογράφους που διδερματίζουν προκειμένου πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ επίσης την προσοχή σας στη σημασία της, στην σημασία της Διεθνούς Επιτροπής για έρευνες. Λοιπόν, να τα διαβάσουμε όλα αυτά πιο προσεκτικά, να δούμε τις στατιστικές. Έχουμε και αποφάσεις δικαστηρίων, μερικές από τις οποίες θα ήθελα να τις αφαιρέσουμε από το κείμενο. Αυτά λοιπόν κλείνω με συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους συνεισηγητές. Ευχαριστώ. Μάιτε Πακατσαουρτούντα. Το, το δοκίμαζα πολλές φορές για να το βγάλω καλά. Και εμείς να επενέσουμε για τη δουλειά που κάνανε οι συνεισηγητές. Άριστη, άριστη δουλειά τους με κάποιες τροπολογίες. Πιστεύω θα πετύχουμε να έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστούμε για την γραμματεία, να μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε αυτή η Επιτροπή. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε και θα πρέπει να επηρεάσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν συνεργάστηκαν όσο περιμέναμε. Και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και την ε, πολιτική υποχρέωση προς τους Ευρωπαίους που έχουν προσδοκίες και να μην υπάρχει συστηματική και συστημική ε, αποφυγή των ε, φορολογικών υποχρεώσεων και διάπραξη όλων των αδικημάτων. Πρόκειται για αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε είναι και εμείς οι ίδιοι να αποκτήσουμε μια σφαιρική γνώση για το τι χρειάζεται το σύστημα για να είναι αποτελεσματικό. Πάρα πολύ καλά τα είπατε κύριε Κόβοντα. Δεν είναι όλοι υπεύθυνοι οι οδηγίες δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε από κάθε όργανο, ε, είτε ήταν αυτό δικαιοδοτικό είτε πολιτικό. Γι' αυτό και λέω να έχουμε μια οπτική όλου του τοπίου και έτσι να μην έχουμε μόνο αντίδραση από συγκεκριμένους. Θα πρέπει να επιστατεύσουμε ό,τι μπορούμε. Και όσο και να προσπαθούν οι διαπράττοντες σε αυτά τα αδικήματα, εμείς θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, χρειάζονται κυρώσεις, ας γίνουν αυστηρότητες. Ούτως ώστε αυτή η ενδιάμεση, οι τράπεζες, όποιος και να είναι, να μην ξανακάνει τα ίδια στο μέλλον. να υπάρξει επίσης ένα νέο κέντρο συντονισμού της ε, φορολογικής πολιτικής και φορολογικής υποπτίας. Άρα έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτά. Όλες αυτές οι συστάσεις που θα διατυπώσουμε να ενεργήσουμε έτσι ούτως ώστε να έχουν καρπούς. Να δούμε επίσης τι παραθυράκια υπάρχουν και όσον αφορά τις, ε, την πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά. Ε, τους ορισμούς να φροντίσουμε, γιατί τώρα πολλά ξεφεύγουν από την τσιμπίδα. Ε, επίσης, να λάβουν υπόψη τα συμπεράσματα της τάξη 1 και συμπαθάτε που ξεπέρασε το χρονικό όριο. Πρόεδρος. Φάμπιο Ντιμάση, εκ μέρους της ΓΟΕ. Ευχαριστώ πολύ τον Γεπεκόφωτ και τον Πέτρο για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε προπερασκευάσοντας ε, τα έγγραφα. Έχουμε παίξει τα 90 λεπτά του αγώνα, έχουμε περάσει πια στην ε, παράταση και πρέπει, γιατί έχει περάσει και η μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο, να ετοιμάσουμε μια καλή ομάδα, μια γερή ομάδα για να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί αυτό θα είναι το κριτήριο το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορέσει να μεταφραστεί σε πολιτική, σε πολιτικές επιλογές. Ένα-δύο σημεία μόνο σε σχέση με την όχι τόσο καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη από πλευρά του Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει συγκεκριμένα να παραπέμψουμε σε οδηγίες που έχουν παρεμποδίσει την διεύρυνση των δικών μας αρμοδιοτήτων από πλευρά της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα έπρεπε να ε, προβλέψουμε ένα σύστημα με το οποίο θα κλητεύονται μάρτυρες, θα ορκίζονται και θα έχουν και τις σχετικές ποινικέ κυρώσεις όταν δεν συνεργάζονται ή δεν ε, τηρούν τον όρκο τους. Ε, οι διαπραγματεύσεις τώρα για την περαιτέρω νομοθεσία, όπως υπόθηκε, έχουν περάσει τον τριμερή διάλογο. Είμαι και εγώ μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο. Πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία να κλείσουν τα παράθυρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τελικό αποδέκτη του ωφέλους. Πρέπει να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Πρέπει να κλείσουν τα παραθυράκια τα σχετικά με τις ε, ε, εταιρείε ε, γραμματοθυρίδες. Και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει περιγραφή του φορολογικού αδικήματος κατά τρόπο που να, επιτρέπει στον ε, εισαγγελέα να ε, διώκει ακόμη και έξω από τα όρια της επικράτειας εάν κάποιος έχει λησμονήσει να δηλώσει ένα σημαντικό πόσο εσόδων. Ο συντονισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως ως προς, την, ε, ως προς τον υπολογισμό στο CCTV της βάσης πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μηδενικό φορολογικό κριτήριο για, τον, ε, για την εγγραφή στη μαύρη λίστα. Βεβαίως, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πρέπει να έχουμε μαύρη λίστα και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε διπλές δυνατότητες φορολόγησης, φορολόγηση βάσεως ε, ε, και άλλωστε έχει προτείνει και η Προεδρία της Μάλτας ότι η φορολόγηση βάσεως ε, θα, είναι, θα πρέπει να είναι ο μοναδικός λόγος εγγραφής στη λίστα. Βέβαια κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θέλουμε φορολογικές κυρώσεις ε, εν ώψη αυτής της μαύρης λίστας. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά. Εμείς ως ομάδα έχουμε κάνει μια ε, μελέτη για τους λεγόμενους enablers, αυτούς δηλαδή που διευκολύνουν την απόκρυψη φορολογικών εσόδων ε, ε, ή, άλλων, ή ε, την απόκρυψη εσόδων. Θα σας διαθέσουμε τα σχετικά κείμενα και τις προτάσεις μας, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έχει τεράστια σημασία το θέμα αυτό και η έκθεση της Europol άλλωστε το είχε επισημάνει και ξέρουμε ότι και η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ Φάμπιο, εκ μέρους των Πρασίνων, η κυρία Χάουταλα. Like to... Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και τη γραμματεία. Εντυπωσιακή η δουλειά που έγινε. Έχω μια-δυο παρατηρήσεις πέραν όσων πει η Μόλι όσον αφορά την ε, πληροφόρηση. Ξανασυναντούμε αυτό το διοργανικό πρόβλημα ε, όσον αφορά το Συμβούλιο. ήταν τροχοπέδι στη δουλειά μας το Συμβούλιο. Δεν μας έδωσαν πληροφορίες. Η Κομισιόν τώρα. Μας έδωσαν πρόσβαση κάποια έγγραφα μόνο σε κάποιο ασφαλές χώρο. αλλά τα περισσότερα από αλλού τα μάθαμε. Ε, αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Δύο ερωτήματα. Τι θα κάνουμε με τα έγγραφα τα οποία έχουν διαβαστεί στην ε, Επιτροπή μας. Αυτό είναι άμεσο. Πρέπει να το λύσουμε. Επίσης, πώς θα εξασφαλιστεί το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες που έχουν τα άλλα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να αντιδραματίσει τον ρόλο του ως ε, ε, ελεγκτικό όργανο. Βεβαίω και θέμα διαφάνεια και προσβασιμότητας πληροφορίες από πλευρά του κόσμου και όχι μόνο από πλευρά του Κοινοβουλίου ω θεσμικό οργάνο. Άρα θα πρέπει αυτό το δικαίωμα του κόσμου να το υπερασπίσουμε. Και τώρα που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα και έτσι οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες γιατί την περασμένη εβδομάδα στην ψηφοφορία περιεστάλλει αυτό το δικαίωμα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην είμαστε υποκριτές. Ίσως αυτό το οποίο έγινε μπορεί να διορθωθεί σε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ Χάγε Χάουταλα. Ο Νούνιο τώρα, ΕΛΚ, και τρεις στο Catch Άννα Γκόμες, Ράμον, Γιουρέγκη, Λουί Μισελ, Τόμας Μαν και ο κύριος Τόιρερ. Παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημασία να βεζόμαστε στα γεγονότα και όχι σε γενικολογίες. Αλλιώς θα πρόκειται για οικοτολογία. Εδώ έχουμε μια έκθεση η οποία επαναλαμβάνω πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα. Να λέει τι μπορεί να βελτιωθεί, τι πρέπει να βελτιωθεί. Ώστε η έκθεση να είναι αξιοποιήσιμη. Τότε θα έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας. Μην ξεχνάτε την εντολή της Επιτροπής μας. Έχουμε ένα στόχο. Αυτό καθορίζεται πάντα. Να συντάξουμε λοιπόν μια έκθεση η οποία θα αντικατοπτρίζει αυτόν τον στόχο και θα τον υπηρετεί. Έχει επίση μεγάλη σημασία να τονίσουμε ποιοι συνεργάστηκαν και ποιοι όχι, ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να έχουν συνεργαστεί περισσότερο, ή ποιοι αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίε. Δείτε τι γίνεται στον τύπο στην κάθε χώρα. Πολλοί μίλησαν στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μίλησαν με εμά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το θυμόμαστε παρακαλώ στο μέλλον. Να θυμόμαστε λοιπόν ποιοι συνεργάστηκαν και ποιοι όχι. Ναι, βεβαίω θα πρέπει να το συμπληρώσουμε και αυτό συγκεκριμένε ε, έρευνε ε, που γίνονται σε σχέση με τα κράτη-μέλη και ή ε, που θα πρέπει να λάβουμε από συγκεκριμένου ε, ιδιώτες, από φυσικά πρόσωπα. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστήσω συνεισηγητές και γραμματεία. Έξοχη δουλειά. Το κείμενο είναι εύληπτο, κατανοητό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι ως κοινοβούλιο. Πέραν των άλλων όμως στόχων κλπ. Νομίζω ότι μπορούμε βραχυπρόθεσμα να επηρεάσουμε τα πράγματα με τον εξή τρόπο, με την έκθεσή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορούμε να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την πέμπτη οδηγία κρατού ξεπλήματος με την οποία θα κλείσει η Εστονική Προεδρία. θέλω να ενημερώσουμε τους ε, εμπλεκομένους, να τους γνωστοποιήσουμε τα συμπεράσματά μας και να επηρεάσουμε παραλαμβάνω την διαπραγμάτευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλήθεια, γιατί ξέρετε, όταν δίνουμε έναν αγώνα δεν είναι μόνο για τη διαφάνεια, για την ισότητα του νόμου, του φορολογικού νόμου, αλλά είναι και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και της τρομοκρατίας. Αυτό το ξεχνούν πολλές φορές τα κράτη μας. Και το λέω αυτό και πάλι εν ώψη της διαπραγμάτευσης περί την πέμπτη οδηγία. Βλέπω τις χώρες μας να μην μπορούν να συμφωνήσουν στην συμπερίληψη των ε, καταπιστευμάτων, των, των trust στην οδηγία. Τέτοιου είδου λοιπόν οντότητε ε, θα διαφύγουν. Πού πάει η διαφάνεια αν δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό δικαιούχο. Επίσης, είναι επίσης σημαντικό το κεφάλαιο περί διευκολυντών, των enablers και περί κυρώσεων. Πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό. Κοιτάξτε, το σύστημα κατά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ. Βασίζεται στην αρχή ότι υπάρχουν υπόχρεες αρχές. Και εμείς εδώ συμπεραίνουμε δυστυχώς ότι τα περισσότερα τέτοια ιδρύματα, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά κλπ. δεν κάνουν τη δουλειά τους τόσο απλά. Κακοδίκηση λοιπόν από κράτη-μέλη αυτό είναι πολύ σημαντικό συμπέρασμα, να το πούμε. Να το γράψουμε στο κείμενο. Και δει στα παραρτήματα και να το αναφέρουμε αυτό και στο πλαίσιο της έκθεσης περί των αποστολών και επισκέψεων σε διάφορες χώρες, όπως στην Πορτογαλία, τη χώρα μου. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες και εξουσίες των διερευνητικών επιτροπών είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να θεσπίσουμε και έναν, διαχωνισμ... και έναν μηχανισμό, με συγχωρείτε, περαιτέρω παρακολούθησης. Γιατί, ωραία, καλοί καταγγέλλοντες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μετά από εκεί. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω ότι περιοριζόμαστε στα δύο λεπτά παρέμβασης. Ραμών, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την έκθεση. Έχω κάποιες νέες παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τη φιλοσοφία του εγγραφού. Εγώ είμαι υπέρ του να επιδείξουμε φιλοδοξία. Δεν συντάσσουμε ε, τώρα ένα νομοθέτημα, έναν χαρτί πορείας, μια μεγάλη διαδρομή, μια πορεία όσον αφορά το να προωθηθούν αυτές οι ιδέες. Αλλά πολλοί κόσμος προσβλέπει σε μας και οπότε θα πρέπει να έχουμε πνεύμα φιλόδοξο και επίσης να έχουμε οριοθετήσει το μέχρι που θέλαμε να φτάσουμε. Θέλουμε επομένω να υπάρχει ένα διεθνές όργανο, οργανισμός, ούτω ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το τι γίνεται όσον αφορά την φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν θέλουμε αυτό να είναι όμως το τέλος. Ε, λέμε για μια επιτροπή για ειδικού του ΟΗΕ, του ΔΕΛΤΑ όμως θα πρέπει συγκεκριμένα να καταλήγουμε σε έναν διεθνή φορέα και έχει να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η συνέχιση και να μην μείνω στο χρονοτούλαπο ε, τα όσα έφτιαξε η τάξη 1, η τάξη 2 και η δική μας επιτροπή θα πρέπει να ε, έχουν, έχει η επιτροπή περισσότερες αρμοδιότητες είπαμε ότι δεν έχει νομική δυνατότητα παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Το είπαμε σε επιτροπέ μα. Και επίση, εάν χρειάζεται, α και οι συνθήκε. Και έτσι να έχει την εξουσία του συντονισμού των φορολογικών και σε, σε με διεθνή οδέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει αυτό να το πούμε. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε πώς θα είναι πιο σαφής η έννοια του αφέμητου ανταγωνισμού διότι πίσω από αυτήν την έννοια έχουμε κάποιο είδους πολύ αθέμητες πρακτικές και αφορούν τα κράτη. Να δούμε επομένω τι είναι θεμητός και τι αθέμητος συναγωνισμός. Στην άποψη ξέρω ότι έχουν λάβει κάποια έκθεση όσον αφορά τις ερευνητικέ επιτροπές και η εμπειρία είναι σημαντική που θα αποκομίσουμε και να καταλήξουμε ο κανονισμός τελικά του Κοινοβουλίου να προβλέπει σημαντικές αρμοδιότητες ερευνητικές. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο θα πρέπει να το συστήσουμε το σημείο αυτό. Ο Λουί Μισελ τώρα, Άλντε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε συνεισηγητές και γραμματεία. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τι θα βάλουμε στις συστάσεις αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό πρέπει να είναι στόχος, ο κύριος στόχος μας. Εν παρόδο, διακρίνω τη συνεργασία με την Κομισιόν από αυτήν με το Συμβούλιο. Η Κομισιόν ήταν πιο δραστήρια, μας βοήθησε, ήταν πιο ανοιχτή. Πραγματικά βοήθησε. Το Συμβούλιο είναι άλλη ιστορία. Για το σύνδεσμο μέλο. Έχουμε εντολή, ναι να υλοποιήσουμε την εντολή. Ας μην αναλωθούμε σε περιφερειακά ζητήματα. Κυρώσει, εργασία, πληροφορία κλπ. Αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επίση για τις συστάσεις χωρίς να αλλάξουμε φυσικά τις συνθήκες. Έχουμε ευθύνη, αλλά πολιτική ευθύνη έχουν τα κράτη-μέλη. Και αυτά πρέπει να ασχοληθούν από εκεί πέρα με την τροποποίηση των συνθήκων. Ε, ίσως πρόεδρε να θεσπίσουμε ένα ελάχιστο ποσοστό αλλά και ένα μέγιστο. Αν έχουμε το ένα πρέπει να έχουμε και το άλλο. Αλλά δεν ξέρω τι είδους εργαλείο θα ήταν αυτό. Και τελευταία παρατήρηση, δεν είμαι υπέρ του να επιδοθούμε σε έναν αγώνα θέσπισης μηχανισμών ελέγχου. Α δούμε τα όρανα που έχουμε στα χέρια μας, τους μηχανισμούς που έχουμε στα χέρια μας, ποια πρέπει να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε τις θερμοδιαιτητέ τους. Α βελτιώσουμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας και μετά ίσως ας αρχίσουμε να ιδρύουμε και άλλου μηχανισμούς, διαδικασίε κλπ. Έχουμε τα μέσα. Ας τα βελτιώσουμε. Έλεγχο χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ω θέμα συζήτηση αυτό του ελάχιστου και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή. Αλλά το έχουμε ξαναδεί ε, με τον ΦΠΑ όπου μείναμε στο 15% για ελάχιστο συντελεστή ε, με βέβαια εξαιρέσεις προβλεπόμενες και ε, με απόλυτη αποτυχία ως προς τον προσδοσμό ανώτατου συντελεστή. Το μας ε, για τους συναδέλφους ε, συνεισηγητές θέλω να πω ότι λυπάμαι αλλά μόνο επένους ακούτε σήμερα και δυστυχώς και εγώ δεν μπορώ να διαφύγω από αυτή τη γραμμή εξαιρετική ήταν η δουλειά που κάνατε και καθίσατε ε, με την έκθεση σας σαφές γιατί έγινε αυτή η διερευνητική επιτροπή και όχι μια έκτακτη επιτροπή, μια ειδική επιτροπή και επίσης βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι με, την, ε, με τις επισκέψεις και τις αποστολές σας μάθατε πολλά πράγματα, πράγματα και μάλιστα πήγατε ενημερωμένοι προκαταβολικά στις ε, χώρες που επισκεφθήκατε. Ξέρατε τι θέλατε να ρωτήσατε και κάνατε τις δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Διερευνητική Επιτροπή. Ξέρουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως λησμονείται σε ορισμένες ε, χώρες. Αν ε, που παραπέμπει στην οδηγία για την καταπολέμηση νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Θέλω να επισημάνω το εξή, ότι η φορολογική αυτή παράδειση θα πρέπει να ξεφωνιστούν, θα πρέπει να κάνουμε έναν κατάλογο και να πούμε πρέπει να, βοηθήσουν τα κράτη, να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά τα οποία ε, έχουν κάνει μια προσπάθεια για να ξεκαθαρίσουν το φορολογικό τους τοπίο και στα άλλα τα οποία δεν ε, έχουν αλλάξει συμπεριφορά να επιβάλλονται κυρώσεις αυτά που θα είναι στη μαύρη λίστα. Για την ε, νομοποίηση παρανόμων εσόδων είναι ένα φαινόμενο πρέπει να πούμε που δεν εκδηλώνεται μόνο σε τρίτα κράτη, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι πιο επικοδομητική βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο το να θεωρούμε ότι θα κάνουμε τροποποίηση τη νομοθεσία ε, νομίζω ότι θα μα καθυστερήσει πάρα πολύ. Και βεβαίω βεβαίως, ε, δεν έχω παρά να διαμαρτυρηθώ για το πόσο καλή είναι η δουλειά που κάνανε οι δύο συνεισηγητέ. Πρόκειται για μια ε, επιτροπή η οποία έχει συνεισφέρει τα μάλα στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Μασμάν. Κύριο Στόιρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερο τους δύο συνεισηγητές. Είναι πολύ καλή έκθεση. Στηρίζεται και στα απορίσματα των δύο ειδικών επιτροπών, τάξη 1 και τάξη 2. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι μια Εξεταστική Επιτροπή και δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Τόμας Μαν ότι έχει άλλα καθήκοντα η ε, Διερευνητική Επιτροπή από την Ειδική Επιτροπή. Ε, είχαμε τον Μάριου Σκόλα από το Λουξεμβούργο που ήρθε στην Επιτροπή τάξη 1, τάξη 2 στις ακροάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Μέχρι σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή δεν κατάφερε να φέρει τον κύριο Μάριου Σκόλ, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο ρόλο διαδραματίσει ως προς τις φορολογικές ε, προκαταρκτικές συμφωνίες του Λουξεμβούργου, ενώ νομίζω ότι ε, τα έγγραφα τα οποία είχαν ζητήσει δύο επιτροπές τάξη 1, τάξη 2 ακόμα δεν έχουν κατεθεί στο Κοινοβούλιο είναι ζήτημα των αρμοδιοτήτων ε, των διερευνητικών επιτροπών και πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη δουλειά επιτελέσει η δική μας Επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε και να υποτιμούμε τις ε, προσπάθειες και το αποτέλεσμα του έργου των ε, τάξε 1 και τάξε 2, των δύο αυτών προ, ε, κατόχων ούτως υπήν. Έγινε μια συστηματική ανάλυση Βεβαίω είχαμε τον περιορισμό με την τάξη 1 και τάξη 2 ότι δεν μπορούσαμε να διερευνήσουμε ει βάθο ορισμένα σημεία και θεωρήσαμε ότι με την Διερευνητική Επιτροπή, την Πάναμα, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προχωρήσαμε όντω περισσότερο από ό,τι πριν, αλλά δεν φτάσαμε ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε. Θα χρειαστεί πολύ ακόμη χρόνο ώστε να πείσουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει να καταθέσει ενώπιόν μας. Βέβαια το ζήτημα είναι αν και η πολιτική ευθύνη για ένα επιθετικό φορολογικό σύστημα έχει καλυφθεί επαρκώς εν ώψη και της ε, Προεδρίας της Μάλτας ε, και των θέσεων του Πρωθυπουργού της Μάλτας εμένω σε αυτά που είπα. Εάν ε, μέλος κυβέρνησης εμπλέκεται σε θέματα που το φέρνουν να ε, μαρτυρήσει ή το, μας οδηγούν να το καλέσουμε να μαρτυρήσει ενώπιον, να δώσει μαρτυρία ενώπιον της Επιτροπής ε, για τα έγγραφα του Παναμά, θα πρέπει να γίνεται αυτό FIU, η Financial Intelligence Unit, δεν μα έδωσε τα στοιχεία που περιμέναμε, αλλά και η επίσκεψη στη Μάλτα δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί όπω θέλαμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει το θέμα τη διερευνητική επιτροπή, καλύτερα τη εξεταστική επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το επαναφέρουμε στην επικαιρότητα. Θα χρειαστεί βέβαια αναθεώρηση των συνθήκων, θα χρειαστεί οπωσδήποτε και υποστήριξη των εθνικών κοινοβουλίων στην ε, υπόθεση αυτή και εδώ νομίζω ότι έχουμε το ε, την κύρια δυναμία, γιατί δεν μας έχουν υποστηρίξει επαρκώς τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι το συμπέρασμα, Πρόεδρο, ότι δεν έχουμε νομοθετικές μόνο ελλείψεις, νομοθετικά κενά ή παραθυράκια, αλλά και κενά εκτέλεσης Εφαρμογή τη νομοθεσία και σε αυτό χρειάζεται σοβαρή αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ Μιχέλ Τόιρερ. Δεν ε, καλούμαστε εδώ να αξιολογήσουμε ποια επιτροπή έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι, το, ότι οι εξουσίε σχετικέ με τη διερεύνηση προβλημάτων ή σκανδάλων τέτοιων δεν έχουν διαμορφωθεί κατά επαρκή τρόπο και στην υπόθεση των τάξε 1 και τάξε 2, αν πρέπει να πούμε τα ονόματα Ναομάριου Σκόλ και άλλοι, αρνήθηκαν να προσέλθουν όποιον τη Επιτροπής. Το Συμβούλιο διατύπωσε σύσταση ε, για αυτοσυγκράτηση. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου διατύπωσε μια πραγματογνωμοσύνη μεταξύ εξαναγκασμού και ε, αυτοσυγκράτηση, ήταν κάπω ανάμεικτη δηλαδή η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε τη δουλειά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα να σα πω κάτι. Το οποίο συνεχίζει με κάποιοι συνάδελφοι, να πω πρώτα-πρώτα ότι αναγνωρίζω το έργο των συναδέλφων, αυτό το σχέδιο κειμένο το οποίο είναι πάρα πολύ σωστή αφετηρία για τη δουλειά τη Εθνική Επιτροπής μα Πρώτα-πρώτα ε, λέγεται στο κείμενο ότι θα πρέπει εγγράφος να αναγνωριστεί και έτσι αυτό να είναι αποδοτικό. Ποια είναι τα όρια μια ερευνητική επιτροπή του Κοινοβουλίου. Αυτό πάρα πολλέ φορέ είναι δύσκολο να το ρεφετήσει κανεί γιατί ε, έχουμε εδώ πέρα διάφορες προσκλήσεις, έχουμε διάφορες ακροάσεις, τη μία μετά την άλλη στην Ερευνητική Επιτροπή. Όμως το σημαντικό ποιο είναι. Θα πρέπει εγγράφως να διατυπώνονται ε, όλα αυτά στα οποία καταλήγουμε ούτως ώστε να χαραχτεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της ε, φοροδιαφυγής, κατά της φοροφυγής και των παραδείσων και θα πρέπει επομένως έτσι ο στόχος να καθοριστεί καλύτερα. Αλλιώς, αλλιώς όλα αυτά υποβιβάζονται όσον αφορά τη σημασία τους και η φορολογική παράδοση και όσον αφορά τις αθέμιτες φορολογικές πρακτικές και στρατηγικές γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιόμορφες ε, καταστάσεις και πολιτικές είδατε τι με τα ελεύθερα λιμάνια τους, τις ζώνες ε, ε, χαμηλής φορολογίας ο στόχος είναι από πλευράς μας να σταματήσει η ατιμορρυσία για την μαζική φοροαποφυγή. Να, περί τίνος πρόκειται τώρα για τα πάνω μαλλίξια, και για τις ε, αποκαλύψεις και βλέπετε πόσες είναι οι χώρες που δεν συνεργάζονται αυτή η φορολογική παράδοση παράδειση και πολλές φορές αυτή η φορολογική παράδοση συνδέονται με τα κράτη-μέλη πούμε αυτές οι υπερπόντιες κτίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή κάποιοι νήσοι της Καραϊβικής που θεωρείται ότι έχουν στρατηγική αξία, μηντική αξία για τις κάτω χώρες. Άρα προσοχή να μην ε, απονευρώσουμε, να μην, να μην υποβαθμίσουμε τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Άρα θα πρέπει να μπορέσουμε ε, σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο θα πλευράς ε, συνδικών να αναβαθμιστεί η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε τι θα γίνει με τα tax rulings για ε, και όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω εξαντλήσαμε την, ε, τις τοποθετήσεις από πλευράς των ε, βουλευτών. Θα παρακαλέσω τους δύο συνεισηγητές να απαντήσουν έκαστος από πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Σκόφωτ. Ευχαριστώ. Σας, τους συναδέλφους, Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αν έχετε και άλλες προτάσεις συγκεκριμένες, ευχαρίστως, θα τις ακούσουμε. Τώρα, να πω δύο λόγια για δύο θέματα. Η Επιτροπή μας, η Πάνα, όντως το είπατε μερικοί από εσάς, ότι είναι μια διερευνητική επιτροπή με περιορισμένες αρμοδιότητες. Αυτό το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό υποβάλλουμε προτάσεις για άλλες επιτροπές και το Κοινοβούλιο εν γέννη. Όμως η φύση του έργου μας είναι να διεισδύσουμε στα γεγονότα, να εξηγήσουμε την φοροποφυγή και φοροδιαφυγή, τη σύνδεση με εγκληματικές δραστηριότητες, να αναδείξουμε τον ρόλο των ενδιαμέσων, των διευκολυντών κλπ. Ας πούμε, η Βρετανική επικράτεια και άλλες επικράτειες εξυπηρετούν διάφορους τέτοιους παράξενους ενδιαμέσους. Θέλησαμε λοιπόν να παρακινήσουμε σε δράση. Ο στόχος μας, το είπαν και πολλοί από εσάς, είναι να δείξουμε στους πολίτες μας, στα κρατημέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πραγματικά ανάγκη να κάνουμε κάτι για το θέμα. Για κάποια επιμέρους πιο συγκεκριμένα θέματα, να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι φανερό νομίζω ότι οι διάμεσοι δικηγόροι, επενδυτές, ε, φοροτεχνικοί κλπ. Τα αυτορυθμιζόμενα επαγγέλματα δεν κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Εδώ έχουμε σημαντικέ ελλείψει. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και ο συνάδελφος Νίντερμάιερ. ναι, έχετε δίκιο. Δείτε τι γίνεται και με τα Panama Papers. Ε, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, όμω εν γέννη το θέμα είναι ότι όταν δεν καταγγέλλονται οι περιπτώσεις αυτές, το πράγμα συνεχίζει οι ενδιάμεσοι αυτοί συνεχίζουν ανενόχλητοι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διαφάνεια. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και ειλικρινή συνεργασία. Όσον αφορά λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, ναι να το δούμε, αλλά να μην ξεχνούμε ότι ο βασικός στόχος είναι η διαφάνεια. Τώρα για την εξωτερική και εσωτερική διάσταση. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά παραθυράκια που διευκολύνουν φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Τα μελετήσαμε αυτά πολύ προσεκτικά. Ε, πρέπει να τα κλείσουμε αυτά τα παραθυράκια με την νομοθεσία μα Τεράστιο έργο για τι χώρε μέλη και την Κομισιόν. Η Κομισιόν να κοιτάξει να κάνει τι μπορεί να κάνει σε εθνικό επίπεδο. Τώρα όσον αφορά τι τρίτε χώρε, κάποιε ε, δεν συνεργάζονται, άλλε είναι υψηλού κινδύνου. Εκεί για να αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να θεσπίσουμε κυρώσει εάν κάποιοι δεν τηρούν τα πρότυπα που έχουμε συνομολογήσει. Για τον πραγματικό δικαιούχο, πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά και τα Panama Papers. Και εκεί κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί, ενώ και τις πέμπτες οδηγίες. Χρειαζόμαστε όμως δράση σε ενωσιακό επίπεδο. Για την εταιρική φορολογία και τον κώδικα δεντολογίας. Χρειαζόμαστε μια συνολική αξιολόγηση του έργου, μάλλον τη απόδοση αυτού του κώδικα, ο οποίο υπάρχει εδώ και 9 χρόνια. Και υποτίθεται ότι χάρη σε αυτόν θα καταργηθούν η φορολογική παράδοση, Και με συγχωρείτε. Κι όμως υπάρχει τόση μυστικότητα, τόση ανωνυμία, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Κομισιόν πρέπει να κάνει τη δική της αξιολόγηση. Έχει αρμοδιότητα να το κάνει, έχει εξουσίες και αρμοδιότητες. Θα την υποστηρίξουμε στην προσπάθεια επίτευξης περισσότερης διαφάνειας και βελτίωσης του κώδικα για την εταιρική φορολογία. Ακούσαμε επίσης πολλά για τις φυστάμενες νομοθεσίες, τις αλλαγές που πρέπει να επιδιώξουμε ναι, ε, αν θέλετε να μιλήσουμε για την κοινή ενωπημένη βάση φορολογία εταιριών, ε, θα αξιοποιήσουμε και εκεί τα ευρήματά μα, όπω είπε ο Ραμόν και άλλοι. Επειδή δεν είναι μια έκθεση νομοθετικού περιεχομένου, είναι απλώ αποτέλεσμα μια διερεύνησης, εδώ πρέπει να είμαστε αυστηροί, πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και φιλόδοξοι και να δείξουμε το δρόμο προ ένα φορολογικό, ένα νομικό μάλλον σύστημα που θα ικανοποιεί τι ανάγκε του 21ου αιώνα. Το σημερινό δεν επαρκεί. Και κανεί δεν έχει την πολυτέλεια να μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Α αλλάξουμε λοιπόν την σημερινή κατάσταση. Σταματώ εδώ πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σα ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Τα σημείωσα. Θα συνεργαστούμε και όσον αφορά τις τροπολογίες και θα καταλήξουμε σίγουρος σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο. Πίτερ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω Στο όσα μόλις ακούσαμε. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Κυρίως για τα θετικά, αλλά όχι μόνο για τα θετικά σχόλια. Να θυμίσω την προσέγγιση μας με την ευκαιρία. Δεν θελήσαμε να υιοθετήσουμε μια ιδεολογική προσέγγιση. Ξέρετε, τα συμπεράσματα βασίζονται στα ευρήματά μας, τα κοινά ευρήματα. Τα συμπεράσματα μετά μεταφράστηκαν σε συστάσεις, όπως γνωρίζετε. Ελπίζω κατά τα άλλα η συζήτηση να οδηγήσει σε τροπολογίες που θα αντικατοπτερίζουν αυτήν την προσέγγιση. Και όλα αυτά ελπίζω να τεκμηριωθούν από τα ευρήματά μας. Μόνον εφόσον η τελική έκθεση, το τελικό κείμενο είναι αξιόπιστο, τότε μόνο θα το πάρουν όλοι σοβαρά και θα συμβάλλει στη βελτίωση του έργου στο μέλλον παρομοίων επιτροπών, επιτροπών διερεύνησης. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ αν και με ελάχιστο προσωπικό, αυτό δεν το θεωρώ κακοδιοίκηση, αλλά έτσι δουλεύει το σύστημα των επιτροπών διερεύνησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχές του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Να είστε σίγουροι ότι συμβάλλετε στην καταπολέμηση της φοροποφυγής, φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος αλλά δείχνεται και το δρόμο για παρομοίες επιτροπές στο μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ όλους όσοι σήμερα τοποθετήθηκαν, ιδιαίτερα τους δύο συνεισηγητές. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική βάση για περαιτέρω δουλειά για μας. Η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογίων ορίζεται για τις 5 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι, πρόκειται για ημέρα Τρίτη. Έχουμε και την εβδομάδα των επιτροπών στη συνέχεια, στην οποία θα μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση των διαφόρων τροπολογιών. Ξεκινούμε τους ή άλλως ε, και με την περίοδο αυτή των διακοπών. Ευχαριστώ ρητά και εγώ την ε, γραμματεία για την ε, πολύ καλή συνεργασία στην προετοιμασία και θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ότι αύριο στις 2 έχουμε τέσσερις υπουργούς των οικονομικών παρόντες. Παρακαλώ να είμαστε στο δυνατόν περισσότεροι παρόντες. Ξέρω ότι, και αύριο, ότι αύριο συμπίπτουμε με συνεδριάσεις επιτροπών άλλων κτλ. Αλλά είπαμε ότι έχουμε τους υπουργούς των οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, των κάτω χωρών, της Ιρλανδίας και αποτελεί η παρουσία τους μια πολύ καλή βάση για ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια έχουμε το, τις διακοπές ε, μετά την κατάθεση των, μετά την προθεσμία για την κατάθεση ε, των τροπολογιών έχουμε το ε, τη συνεδρία της 26 Σεπτεμβρίου με ένα θέμα το Football Leaks και ένα θέμα διαμόρφωση φορολογικών διευκολύνθησεων <coughs> MSF και Caterpillar. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά να είστε όσο το δυνατόν περισσότεροι αύριο. Όσοι όμως δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αν και ελπίζω να είναι ελάχιστοι, εύχομαι να έχετε πολύ καλές διακοπές. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και οι διερμηνείς ευχαριστούν.